Good. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω όλους θερμότατα και κηρύσω την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής μας. Το πρώτο θέμα είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης λόγω του γεγονότος ότι από ό,τι φαίνεται έχουν να συζητήσουν πολλά οι συντονιστές θα σας πρότεινα την εξής αλλαγή στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Προτείνω λοιπόν τα σημεία 5, 6 και 7 να αναβληθούν συγκεκριμένα το 5 και το 7 για το αμέσως επόμενο διάστημα, το νωρίτερο δυνατό, ενώ το 6 αύριο το πρωί πριν τις ψηφοφορίες να το συζητήσουμε, διότι πρόκειται για την έκθεση που έχει σχέση με την επικουρικότητα, όπως ξέρετε. Επαναλαμβάνω, το σημείο 5 και 7 αναβάλλονται για επόμενη συνεδρίαση, όσο γίνεται πιο γρήγορα βέβαια, ε, και αύριο το πρωί να εξετάσουμε το σημείο 6 πρώτο πριν τη ψηφοφορία. Εντάξει. Οπότε θα μπορούσε στις 4.30 να αρχίσει η συνεδρίαση των συντονιστών για να έχουμε χρόνο ενδιάμεσα να συνεννοηθούμε και να κανονίσουμε. Γιατί έχουν πολλά θέματα στους συντονιστές. Συμφωνείτε με αυτή την πρόταση, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα να μάθω για ποιο λόγο το ζητάτε αυτό, για ποιο λόγο αναβάλλονται αυτά. Ε, δεν μας δώσατε το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να υποστηρίξω ρητά την πρόταση, λέει ο κύριος Κασπάρη. Στις δύο τελευταίες συνόδους Ολομέλειας από την Επιτροπή μας δεν δώσαμε την καλύτερη εικόνα. Είχαμε ένα θέμα στο οποίο είχαμε επίμαχη ψηφοφορία ε, για τα μεταλλεύματα από ε, περιοχές εμπόλεμη σύρεξη. Ε, η πολιτική μάχη και οι διαπλεκτισμοί κάνουν καλό στη δημοκρατία, αλλά κανονικά αυτά τα θέματα τα συζητούσαμε τα τελευταία δέκα χρόνια στην Επιτροπή πριν φτάσουν στην Ολομέλεια. Και ενώ μια έκθεση είχε ψηφιστεί με τα δύο τρίτα στην Επιτροπή μας, τελικά αφαιρέθηκε από τη μέρηση διάταξη της Ολομέλειας και επαναπέφθηκε στην Επιτροπή μας. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε στο μέλλον πώς θα λειτουργήσουμε, πώς θα συνεννοούμαστε και πώς θα ε, εργαζόμαστε. Γι' αυτό θέλαμε χρόνο ε, στη συνεδρίαση των συντονιστών περισσότερο για να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτά είναι ε, πράγματα ε, που χειρίζεται ο κύριος Σόλτς, ο οποίος μόλις βγήκε έξω, που είναι συντονιστής της ομάδας μου και αρμόδιος για θέματα ενεργειακής ένωσης και δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω τη γνώμη της ΓΚΟΕ. Να περιμένουμε λίγο τον κύριο Σόλτς, δεν μπορώ να σας πω εγώ να δεσμευτώ αυτή τη στιγμή. Καλώς. Αν δεν θέλει κανείς ε, άλλο το λόγο, έτσι λοιπόν θα προχωρήσουμε. Επαναλαμβάνω, τα σημεία 5 και 7 αναβάλλονται. Με τον κύριο Μπούχνερ να δούμε μήπως μπορούμε να το συζητήσουμε αύριο το απόγευμα και το θέμα της κυρίας Σάκε ε, θα το κανονίσουμε για άλλη φορά. Το σημείο 6 θα συζητηθεί πρώτο αύριο το πρωί στις 9 πριν τις ψηφοφορίες διότι πρέπει και να ψηφιστεί. Και η συνεδρίαση των συντονιστών θα αρχίσει στις 4.30. Damit stelle ich die Tagesordnung... Λοιπόν, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη ούτως τροποποιηθήσα. Ε, ερχόμαστε στο δεύτερο θέμα, έγκριση των πρακτικών. Όπως πάντα... Α, ο Γιάννικ ε, Ζαντό. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην ημερήσια διάταξη αύριο το τελευταίο σημείο είναι το FLECT. Το είχα ζητήσει εγώ, έχω δουλέψει πολύ επ' αυτού, αλλά δεν μπορώ να είμαι αύριο παρόν. Ε, μια και δεν είναι επίγον, θα μπορούσαμε να το αναβάλουμε στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε. Οπότε θα έχουμε και περισσότερο περιθώριο κερδίσει για την Ενεργειακή Ένωση και να το συζητήσουμε με μεγαλύτερη ευχέρεια ως σημείο 20 λοιπόν αύριο γιατί θα έχουν φύγει τα δάση και τα λοιπά το φλεκτ. Ωραία. Για τα πρακτικά. Έχετε στα χέρια σας τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης και αν δεν διαφωνήσει κανείς θα θεωρηθούν εγκεκριμένα τα πρακτικά. Σημείο 3. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Όπως πάντα μεταδίδεται απευθείας ε, στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μας και εικόνα και ήχο. Προσέχετε λοιπόν όταν παίρνετε το λόγο και ε, τις κινήσεις σας όλα τα παρακολουθούν πολλοί τηλεθεατές και ακροατές σε πολλές χώρες αυτής της γης. Θα βρείτε ένα κατάλογο της αλληλογραφίας που είχαμε στο φακελό σας. Εάν θέλετε να πάρετε τις επιστολές αυτές, απευθυνθείτε παρακαλώ στη γραμματεία. Ξέρετε ότι έχουμε ακρόαση σήμερα στρογγυλής τραπέζης για τις εξαγωγικές πιστώσεις και αύριο έχουμε ε, μια συζήτηση και στις 17 Ιουνίου για τη διτή χρήση και τον εξυγχρονισμό, το, περίμενο, το περίφημο dual use. Γνωρίζετε ότι φαίνεται να κινούνται τα πράγματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ιαπωνίας. Η τελευταία μεγάλη δραστηριότητα ήταν η εξής το, η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιαπωνίας φαίνεται ε, τέλη του έτους να ε, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και να μπορεί να συνευθεί η συμφωνία με την Ιαπωνία. Ξέρετε ότι στις 18 και 19 του μηνός θα μεταβεί στο Μιλάνο αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας για να ασχοληθεί με την ασφάλεια τροφίμων και την βιωσιμότητα στο παγκόσμιο εμπόριο. Για να ρίξουμε και μια ματιά στην έκθεση του Μιλάνου. Ξέρετε και μάθατε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, έχει οδηγηθεί σε εμπλοκή ε, στη Βουλή των Αντιπροσώπων Οργανισμός Προώθησης Εμπορίου την Παρασκευή ενέκριναν τη συμφωνία με ψήφους 219 υπέρ 211 ε, κατά. Αλλά ε, για το ε, ε Ταμείο Προσαρμογής για την αντιμετώπιση των εργαζομένων που πλήττονται απερίφθη με μεγάλη διαφορά. 126 υπέρ, 302 κατά. Οπότε Μάλλον θα ξανασυζητηθεί τούτη τη βδομάδα, αλλά με αβέβαιη έκβαση. Και δεν ξέρουμε πότε θα εγκριθεί αυτός, ε, αυτή η αρχή προώθηση εμπορίου ε, Trade Promotion Authority. Ε, ασχολείται πολύ εντατικά και η δική τους Βουλή, όπως βλέπετε, με τα θέματα αυτά του διεθνούς εμπορίου και των συμφωνιών του. Έχει συμφωνηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε, ε, ε, σε βάθος εμπορική συμφωνία με την Τινησία. Ξέρετε ότι έγινε μια μελέτη ε, αντικτύπου και πεδίου εφαρμογής και βολιδοσκόπηση για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις σε ευθέτω χρόνο, που δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός. Τώρα, στον ΠΟΕ, τι γίνεται με τα λεγόμενα πράσινα αγαθά, green goods. Ακούμε ότι υπάρχει κάποια πρόοδος, 4 με 8 Μαΐου στη Γενέβη έγινε μια συζήτηση για τον τροποποιημένο κατάλογο προϊόντων που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται εκεί. Η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί αυτή τη βδομάδα 15 με 19 Ιουνίου. Τελευταία ανακοίνωση. Έχουν γίνει τριμερείς συζητήσεις ε, για την συμφωνία με την Ουκρανία. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ουκρανία και τη Ρωσία. Αυτά είναι τα τρία μέρη ε, σχετικά με τις ενστάσεις και τις αντιρρήσεις που προέβαλε η Ρωσία κατά τη Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας για να λυθούν αυτά τα προβλήματα και ξέρετε ότι ε, όλα αυτά γίνονται σε ένα πολύ ειλικρινές και επικοδομητικό κλίμα σε πολλούς τομείς ε, βρέθηκαν και πρακτικές λύσεις οπότε εγώ πιστεύω ότι μπορεί να τεθεί την 1η Ιανουαρίου του 2016 σε ισχύ η συμφωνία. Βεβαίως η ρωσική πλευρά στις 3 Ιουνίου κατέθεσε νέο έγγραφο που ζητεί νέα συμφωνία, τριμερή αυτή τη φορά, που να συμμετέχουν και οι ίδιοι, σε πολλούς τομείς αυτό, πώς να το πω, υπερσκελίζει ή παραφορτώνει τη συμφωνία με την Ουκρανία και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις έχει και αμφιλεγόμενο περιεχόμενο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε αυτό το αίτημα, ιδιαίτερα διότι η ρωσική πλευρά απαιτούσε να υπάρξει δεσμευτική σχέση μεταξύ της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και της νέας υποτιθέμενης συμφωνίας αυτής της τριμερούς. Εδώ νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σωστά αντέδρασε και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε Κατά την άποψή μου όμως δεν επιτρέπεται να συνάπτουμε συμφωνία εταιρική θέση και συνεργασίας στην οποία να είμαστε αναγκασμένοι να τη δεσμεύουμε και να την εξαρτώμε από μια άλλη συμφωνία τριμερή με ένα τρίτο εταίρο. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις που είχα να σας κάνω. Δεν ζητεί κανείς το λόγο, οπότε μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 4 Έχουμε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τις εξαγωγικές πιστώσεις με δημόσια στήριξη, ενίσχυση των εξαγωγών δηλαδή στα κράτη-μέλη. Γνωρίζετε ότι το θέμα και το εργαλείο είναι αυτό σημαντικό στην εμπορική πολιτική για να ε, ανοίγονται αγορές και ευκαιρίες επιχειρηματικές από την άλλη όμως υπάρχουν και κάποιες απαιτήσει για την προστασία του περιβάλλοντος, την αηφόρο τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΣΑ. Και πάντα συνοδεύουν τις εξαγωγικές ενισχύσεις και πιστώσεις. Wir haben jährlich den Bericht über... Έχουμε ετησίως μια έκθεση για τις εξαγωγικές πιστώσεις για το πώς ε, υπάρχουν διάφορα συστήματα στα κράτη-μέλη και πώς εφαρμόζονται και τα συζητούμε κάθε χρόνο. Για να ασχοληθούμε λοιπόν σήμερα σε βάθος, έχουμε προσκαλέσει μία σειρά εμπειρογνωμόνων για μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης. Θα ήθελα ήδη να παρακαλέσω τους εμπειρογνώμονες να μην μιλήσουν περισσότερο από 9 λεπτά έκαστος. για να μπορέσουμε να έχουμε χρόνο για συζήτηση στη συνέχεια. Καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο David Trisdale, που είναι επικεφαλής ε, του αντιστοίχου τμήματος του ΩΣΑ και να του δώσω αμέσως το λόγο. Έχετε το λόγο κύριε Ντράισδελ. Uh, Ευχαριστώ. Θα σας δώσω μία επισκόπηση της δουλειάς που κάνουμε σε εξαγωγικές πιστώσεις στο Παρίσι, στον ΩΣΑ. Ο ΩΣΑ είναι το Διεθνές Φόρουμ για τις εξαγωγικές πιστώσεις εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Το 1963 είχε δημιουργηθεί μια υποομάδα της ε, ε, Επιτροπής Εμπορίου για τις εξαγωγικές πιστώσεις και τις ε, εγγύησεις πιστώσεων. Μια ομάδα η οποία συνεδριάζει τακτικά και συζητάει τέτοια θέματα πολιτικής στον ΩΣΑ. Ανταλλάσσονται απόψεις για το κατά πόσο είναι συνεπής η πολιτική. Παρακολουθούμε τις δραστηριότητες των μελών. Εξετάζουμε θέματα διαφάνειας και αποκαλύψεων. Η Ισλανδία, ε, κατ' εξαίρεση, είναι μέλος επίσης αυτής της ε, ομάδας. Υπάρχουν τέσσερις τομείς εργασίας, ε, διαφάνεια, ανταλλαγή πληροφοριών ε, για τα προγράμματα και τις συναλλαγές. Υπάρχει η συζήτηση των ε, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ε, ε, συναλλαγών που υποστηρίζονται με επίσημα με εξαγωγικέ πιστώσει, Υπάρχει μια σύσταση του ΩΣΑ για την εφαρμογή τη σύμβαση κατά τη δροδοκίας του. Όταν τα μέλη δηλαδή κάνουν τέτοιε συναλλαγέ, λαμβάνουν υπόψη τι προσπάθειες καταπολέμηση της διαφθοράς και της δροδοκίας στι διεθνείς συναλλαγέ. Και έχουμε και μια συμφωνία για την το βιώσιμο δανεισμό μια προσπάθεια να εξασφαλίσουμε ότι δεν προωθούμε στις ε, χώρες που δανείζονται ε, αβίωτα επίπεδα χρέους. Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια. Όλα τα μέλη μας ε, κοινοποιούν τα νέα προγράμματα εξαγωγικών πιστώσεων. Είναι μια προσπάθεια χαρτογράφησης που κάνουμε, όπου παρακολουθούμε και βλέπουμε τα διάφορα προγράμματα που προωθούν όλοι. Όλοι ξέρουν λοιπόν τα προγράμματα των άλλων. Είναι καλό εργαστήρι για να καταλάβουμε οι μεν τους δε και να δούμε τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Ε, γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών για τις υπάρχουσες και αναδυόμενες πολιτικές και όλες οι συναλλαγές ε, αναγράφονται για να τις παρακολουθούμε. Μιλάμε και για τις εξαγωγικές πιστώσεις και για τη βοήθεια που συνδέεται με το εμπόριο. Στα πλαίσια όλα αυτά της καλής διακυβέρνησης. Κάνουμε μια ευρή ανταλλαγή πληροφοριών ε, μεταξύ μας και μεταξύ ημών και μη μελών, γιατί υπάρχουν όλο και περισσότερες χώρες που έχουν τέτοια επίσημα προγράμματα εξαγωγικών πιστώσεων με δημόσια στήριξη. Για το περιβάλλον, εδώ και 20 χρόνια ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις για να έχουμε μια κοινή προσέγγιση, ούτω ώστε όλα τα μέλη να εφαρμόσουν τι ε, περιβαλλοντικέ κατευθυντήριε γραμμέ στα προγράμματα που υποστηρίζουν. Υπάρχει μια εξέλιξη λοιπόν που τη βλέπετε εδώ από την πρώτη ε, συμφωνία του 2003 που αναθεωρήθηκε το 2007 και το 2012 συνεχεία. Και την περασμένη εβδομάδα συζητήσαμε για να λογοδοτήσουμε στο Συμβούλιο για προτινόμενες συστάσεις, τόσο ώστε να ενισχύσουμε περαιτέρω την κοινή προσέγγιση για το περιβάλλον. Πολύ σύντομα. Εδώ τι κάνουμε για το περιβάλλον. Απαιτούμε από τα μέλη να παρακολουθούν τα προγράμματα ε, στους διάφορους τομείς, να κάνουν μελέτες αντικτύπου για το περιβάλλον και τα κοινωνικά θέματα και να ε, ε, σέβονται τα πρότυπα των χωρών που λαμβάνουν αυτά τα προγράμματα, αλλά και τα διεθνή πρότυπα. Και μερικές φορές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περιβαλλοντική πολιτική. Υπάρχουν υποχρεώσεις εκ των εκ λογοδοσίας, ούτως ώστε να παρακολουθούμε την εφαρμογή αυτών των συμφωνιών. Έχουμε μια συμφωνία για το θέμα της δωροδοκίας, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας. Είναι μια σύσταση ότι όλοι προσπαθούμε όταν γίνεται μια αίτηση, να λαμβάνουμε υπόψη μας ε, το κατά πόσον δεν υπάρχει θέμα ε, διαφθοράς, ε, και κατά πόσον ο ετών ε, βρίσκεται σε αυτόν τον κατάλογο ε, διαγραφής λόγω του ότι έχει πάρει δωροδοκία. Με τη διαφάνεια μειώνουμε τις επιπτώσεις της δωροδοκίας. οι αρχές αυτές, ε, αν πιστεύουν ότι υπάρχει δωροδοκία, ε, ασκούν την ε, ρήτρα δέουσας επιμέλειας και παραπέμπουν το θέμα στις κατάλληλες αρχές για να το διερευνήσουν. Οι ECAs, δηλαδή, Οργανισμοί Εξαγωνικών Πιστώσεων. Επίσης, ε, έχουμε την αρχή ε, ε, βιώσιμου δανεισμού στις χώρες χαμηλού εισοδήματο. Υποστηρίζουμε το πρόγραμμα της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δεν θέλουμε να οδηγήσουμε σε υψηλά επίπεδα χρέου σε χώρες, ιδίως αυτές που, λαμβάνουν, που έχουν μέτρα ανακούφισης χρέους. Ε, έχουμε μια άλλη συμφωνία για τις εξαγωγικές πιστώσεις με δημόσια στήριξη. Είναι μια ξεχωριστή συμφωνία που ξεκίνησε το 1978. Αφορούσε τα μέλη του ECG. Εκεί είχαμε τους πρώτους κανόνες συνένεσης για το ποιο θα ήταν η καλύτερη τρόπη χρηματοδότησης των εξαγωγικών πιστώσεων υπάρχουν νέα ε, συμμετέχοντες, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει. Ε, το θέμα αυτό αφορά τους κανόνες χρηματοδότησης. Έχουμε μια ξεχωριστή συμφωνία τομεακή για την, τον αεροπορικό τομέα, όπου συμμετέχει η Βραζιλία γιατί κατασκευάζει πολλά αεροπλάνα. Η Βραζιλία, συγγνώμη, η Τουρκία και το Ισραήλ επίσης είναι παρατηρητές αυτή τη στιγμή. είναι μια συμφωνία κυρίων, ήπια νομοθεσία, εκτός από το νομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετέχουμε, συνεδριάζουμε τακτικά, έχουμε, ε, συμμετέχουμε σε, και συνεδριάζουμε σε επίπεδο τεχνικών εμπειρογνωμόνων με σκοπό να δημιουργήσουμε ισοτιμία στις επίσημες εξαγωγικές πιστώσεις και στην βοήθεια, την εμπορική βοήθεια. Θέλουμε ε, ε δεν θέλουμε να υπάρχουν επιδοτήσεις και να παρακολουθούν οι επιδοτήσει στο βαθμό που γίνεται το, ε, τη στάση του εμπορίου. Και δεν θέλουμε οι κυβερνήσεις να χρηματοδοτούν τις ε, εξαγωγικές πιστώσεις. Υπάρχει αρκετή διαφάνεια στην ε, όλη διαδικασία που μας επιτρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αν υπάρχουν εμπορικές διαφωνίες σε μία συναλλαγή μπορούν να επιληθούν σε πραγματικό χρόνο, τόσο ώστε να μην στραβλώνει το εμπόριο. Ε, οι τομείς που καλύπτονται αφορούν, ε, αφορούσαν ε, το ελάχιστο επιτόκιο και το περιθώριο, το χρόνο δηλαδή πληρωμής, αλλά τελικά μιλήσαμε για, και για άλλα θέματα, για τα ελάχιστα επιτόκια, την ασυνδεδεμένη βοήθεια, τα ελάχιστα ασφάλιστρα κτλ συμπεριλαμβάνεται στη Συμφωνία του ΠΟΕ για τις ε, επιδοτήσεις στο σημείο K που προβλέπει ένα ασφαλή λιμένα εάν οι διατάξεις ε, του, της συμφωνίας αυτής, του arrangement, ακολουθούνται. Και είναι ένα ευέλικτο μέσο αυτό το arrangement. Αναθεωρούμε συνέχεια τους όρους, ούτως ώστε να είναι λειτουργικό. Το πεδίο εφαρμογής ε, ε, καλύπτουμε τομεί ε, χρηματοδότησης πάνω από δύο χρόνια. Ε, αφορά το μη στρατιωτικό εξοπλισμό. Ε, αφορά διάφορα επίσης προϊόντα. Είναι ευέλικτο, διαφανές και επιτρέπει ένα... Μας επιτρέπει να μην έχουμε πολλές συγκρούσεις, γιατί επιλύονται οι όποιες διαφορές σε πραγματικό χρόνο. Η βασική διάταξη είναι η διαφάνεια. Αν οποιοδήποτε έχει δια... ερωτήσεις για μια συναλλαγή, τις υποβάλλει σε πραγματικό χρόνο για να επιληθούν ή για να υπάρχει ισοτιμία τουλάχιστον. Υπάρχει πολιτική δέσμευση για την ε, συμφωνία. Ε, εφαρμόζεται γενικά μέσω της νομοθεσίας σε πολλές χώρες, ε, παρότι σε πολλές χώρες είναι ήπια νομοθεσία, με εξαίρεση βέβαια την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι πραγματική νομοθεσία. Ευχαριστώ. Εκτενέστατη περιγραφή και σκόπιση των δραστηριοτήτων του ΟΣΑ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Αντώνιο Τρικάρικο που εργάζεται για μια Ιταλική μη κυβερνητική οργάνωση και σήμερα θα μιλήσει ε, εξ ονόματος του ECA Watch που είναι η διεθνή Εκστρατεία για τι εξαγωγικέ πιστώσει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπω είπατε, εκπροσωπώ την ECA Watch, η οποία είναι ένα δίκτυο, ένα διεθνές δίκτυο με κυβερνητικών οργανώσεων, που ασχολείται με μια σειρά ζητημάτων, το περιβάλλον, την ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα ε, δικαιώματα τα συνδικαλιστικά και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μας δίνεται ευκαιρία να μιλήσουμε στην Επιτροπή Ίντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ζήτημα αυτό. Πιστεύουμε ότι η δημιουργία αυτού του συστήματος έχει βοηθήσει να υπάρξει μεγαλύτερη λογοδεσία και μεγαλύτερη διαφάνεια στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τρόπο με τον οποίο ε, εφαρμόζονται οι εξαγωγικέ πιστώσεις. Ωστόσο, ε, βλέποντας πώς έχει εφαρμοστεί αυτό και πώς μπορεί να ασχεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την εποπτεία του, υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Έχουν εμφανιστεί ζητήματα συνεκτικότητας της πολιτικής και αυτό μας το έχει δείξει η πρόσφατη δήλωση των G7 για τη συζήτηση που συνεχίζεται σε σχέση με την χρήση του άνθρακα και την κλιματική αλλαγή. Κατά την άποψή μας, η βιομηχανία του άνθρακα είναι σημαντική. Ωστόσο, η προστασία του κλίματο από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακόμα σημαντικότερη. Γι' αυτό θα ήθελα να σταθώ σε τρία κρίσιμα ζητήματα ε, από την πλευρά τη δική σα Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα είναι το ζήτημα τη διαφάνεια Κατά την άποψή μας αυτή η διαφάνεια είναι πάρα πολύ σημαντική και διαφέρει η σεβασμός της ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ε- Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι πρώτα απ' όλα στο γεγονός ότι ορισμένοι δωρητές επιμένουν στο να μην δημοσιοποιούν όπως οφείλουν τις διάφορες ε, ε, πληροφορίες, όπως ιδιαίτερα τις στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Αυτό το είδαμε πρόσφατα, για παράδειγμα, στην επέκταση της διόρυγας του Σουέζ, όπου δόθηκαν πιστώσεις από την πλευρά των Ολλανδίας και του Βελγίου, χωρίς να έχει δημοσιοποιηθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και χωρίς να γνωρίζουμε ποιες είναι επιπτώσεις για τις τοπικές κοινωνίες το οποίο σημαίνει ότι η αναρμόνιση θα πρέπει να βελτιώνει τα πράγματα προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω, κατά την άποψή μας. Θα πρέπει να υπάρχει πληροφόρηση από τα κράτη-μέλη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη σειρά της να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έρχομαι τώρα στο ζήτημα των ενδεχομένων υποχρεώσεων, το οποίο ελάχιστα κράτη-μέλη αναφέρουν στις αναφορές που υποβάλλουν στην ε, ε, Επιτροπή το αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο τα κάθε κράτη-μέλη, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα στοιχεία που έχουμε και να γνωρίζουμε τι ρίσκο αντιπροσωπεύουν οι διάφορε υποχρεώσει που αναλαμβάνονται και δεν εμφανίζονται στου ισολογισμού. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα από την Βρετανία. Η UKEF, ο Οργανισμό Εξωτερικών Επιστώσεων, έχει χρησιμοποιήσει μια ειδική, ε, ένα μηχανισμό, μια ειδικό όχημα, το οποίο ονομάζει Τζεύκο, e για να μην εγγράψει στον ισολογισμό τη παραπάνω από 7 δισεκατομμύρια λίρε. Και παρά το γεγονό ότι είναι γνωστή η ύπαρξη στη, αυτού του φορέα και ότι το γνωρίζει και η Γενική Διευθυνσία Εμπορίου, δεν έχει κινήσει τη διαδικασία, ε, για παράδειγμα, κρατικών ενισχύσεων. Ούτε έχει γίνει μια πιο ενδελεχής έρευνα του προβλήματος, που σημαίνει ότι το ζήτημα αυτό ε, θα πρέπει να εξεταστεί πιο ενδελεχώς στην αρμόδια ομάδα εργασίας του Συμβουλίου και να συμφωνηθούν κοινά πρότυπα για τις αναφορές. Ωστόσο υπάρχει και ένα γενικότερο ζήτημα ε, που το είδαμε με την έρευνα που εξήγαμε πρόσφατα για τα ζητήματα της υποστήριξης των ε, ε, προγραμμάτων εξόριξης άνθρακα, που μας δείχνει ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απευθύνεται στα κράτη-μέλη και να αναζητάει ίδια τις πληροφορίες που θα συνοψίζει στην έκθεσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί πρόκειται για δραστηριότητες οι οποίες δεν εμπίπτουν στο διακανονισμό του ΩΣΑ. Αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν μια σειρά διαφορετικών μηχανισμών χρηματοοικονομικών για αυτού του είδους τις επενδύσεις και η πραγματική πολιτική εποπτεία τους είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Και αυτό ίσως επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καταφέρει να περάσει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των διαφορών διαπραγματεύσεων στον ΟΣΑ και διεθνώς. Θα πρέπει λοιπόν η Επιτροπή να διαρευνήσει τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν αυτού του χρηματοοικονομικού μηχανισμού, ε, του μηχανισμού ενίσχυση. Και έρχομαι στο τρίτο θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί και παραθέτω ότι τα κράτη-μέλη παρήχαν τις απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 και 21 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο διακανονισμός όμως του ΟΣΑ δεν είναι συμβατός 100% με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε πολύ σημαντικά ζητήματα ε, μάλιστα, όπως για παράδειγμα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το οποίο σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να έχει δημιουργήσει μια δική της ε, πλήρη μεθοδολογία για την ανάλυση των, ε, του τρόπου με τον οποίο οι εξαγωγικές πιστώσεις έχουν επιπτώσει σε αυτά τα πρότυπα που ε, έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΙΝΤΑ ίδια το 2013 στην εκθεσή της είχε δώσει την εξή σύσταση. Το... Η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για τις εξαγωγικές πιστώσεις και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να συνεργαστούν για να συμφωνήσουν σε μια νέα μεθοδολογία ε, με την οποία θα εξετάζεται κατά πόσον τηρήθηκε το άρθρο 21 και ο τρόπος με τον οποίο η ε, εφαρμογή του διακανονισμού των και των κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΣΑ έγινε με τρόπο συμβατό με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Δυστυχώς γνωρίζουμε ότι αυτή η διαβούλευση δεν έγινε μέχρι στιγμής. Το μόνο που είχαμε ήταν τη συμμετοχή εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών την προηγούμενη εβδομάδα στη Ρήγα, αλλά και αυτοί περιορίστηκαν σε κάποιες αναφορές στη σχέση του άνθρακα με την κλιματική αλλαγή. Επίσης αναφέρεται, έχει αναφερθεί σε αυτή την έκθεση, η σημασία που έχει να λαμβάνονται υπόψη στις συστάσεις του ΟΗΕ και άλλων διεθνών οργανισμών. Αν και γίνεται τέτοια χρήση αυτών των συστάσεων στην πολιτική εξαγωγικών πιστώσεων, αυτό δεν αρκεί για να πούμε ότι γίνεται σεβαστό το άρθρο 21. Και κλείνω λέγοντα ότι μια και την επόμενο μήνα, τον επόμενο μήνα η Επιτροπή σα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξετάσει την ανανέωση των κατεξουσιοδιώτης πράξεων θα έπρεπε κατά την άποψή μου να επιμείνετε και να ζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παίξει το ρόλο της για την εφαρμογή του παρατήματος 1 και τη σωστή λογοδεσία και αναφορά προς εσάς, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί ο Δόκτωρ Ιγκο Γιούγκερ που είναι επικεφαλής ε, του τμήματος και του γραφείου συνδέσμου ε, Χέρμες ε, που εδρεύει στο Βερολίνο και ε, είναι ηγετική παγκοσμίως σε θέματα ε, ασφαλίσεων ε, πιστώσεων. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ. Είναι ο Γερμανικός Οργανισμός Εξαγωγικών Πιστώσεων, ο Ερμής, Χέρμες, ο φορέας στον οποίο εργάζομαι. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω κάποιο πλαίσιο τα έχουν ήδη πει οι προλαλήσαντες. Εγώ θα επιμείνω στα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, στη διαφάνεια και κάποια άλλα ειδικά γερμανικά στοιχεία αν υπάρξει αρκετός χρόνος. Εσείς γνωρίζετε πώς έχει η δομή και ο τρόπος λειτουργίας ενός Εθνικού Οργανισμού Εξαγωγικών Επιστώσεων. Να σας δώσω μερικές παραμέτρους όμως για να καταλάβουμε καλύτερα πώς λειτουργεί ο δικός μας οργανισμός. Όπως είπε και ο David Drysdale του ΟΟΣΑ, υπάρχουν διάφοροι τρόποι υποστήριξης ε, ε, των προσφορών των εξαγωγικών πιστώσεων στην Ευρώπη. Ε, η κάλυψη κυρίως κυριαρχεί. Υπάρχουν και συστήματα πιστώσεων άμεσα, αλλά αυτό είναι ε, μάλλον εξαίρεση. Έχουμε συνήθως μια εμπορική τράπεζα που χρηματοδοτεί τις εξαγωγές μιας εταιρεία ε, που χρειάζεται εξοπλισμό κτλ. και το δάνειο είναι μέσω μακροπρόθεσμο για να προωθηθεί η εξαγωγική δραστηριότητα. Για να γίνουν λοιπόν αυτές οι συμφωνίες, οι εξαγωγείς και οι τράπεζες ε, ζητούν εγγύηση ή κάλυψη από το φορέα πρόθεσης εξαγωγών εξαγωγικών πιστώσεων. Δεν είναι κρατική ενίσχυση αυτό σε καμία περίπτωση, ούτε επιδότηση. Θα πρέπει να πληρώνουν ε, κάποιο τέλος ασφάλιστρα ή ε, εξαγωγής και υπάρχει ένα σύστημα ολόκληρο που ε, κανονικά αυτοχρηματοδοτείται και αυτοσυντηρείται τουλάχιστον μέσο και μακροπρόθεσμα. Δεν υπάρχει σύγκριση του δικού μας φορέα με τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ούτε τράπεζες είμαστε αναπτυξιακές, ούτε αναπτυξιακή βοήθεια χορηγούμε, ούτε χρήματα επενδύουμε. Δεν είμαστε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Είναι μια δραστηριότητα που διέπεται από τη ζήτηση. Δεν επιλέγουμε εμείς τα προγράμματα και τις συναλλαγές που πρέπει να υποστηριχθούν. Η αγορά είναι εκείνη και οι τράπεζες που απευθύνονται σε εμά γιατί θέλουν κάλυψη για τις δικές τους εμπορικές συναλλαγές και δραστηριότητες οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων υποστηρίζουν τις πιστώσεις της εξαγωγικής, όχι το έργο το ίδιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν μπαίνουμε στην ουσία του προγράμματος, στις υπηρεσίες λοιπόν καλύπτουμε και τις εξαγωγικές πιστώσεις. Having said this... Τούν των λεχθέντων, δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα είπε ο David Ράιστελ, οι φορείς ε, πρόθεσης των εξαγωγικών πιστώσεων Ήδη έχουν ε, βρει κοινέ ε, προδιαγραφές για την ορθή διακυβέρνηση. Ακούσαμε αυτή την νομοθεσία για το σύστημα για κατά πολέμηση της δωροδοκίας και την ε, αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων με τη δέουσα επιμέλεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ΩΣΑ, το ακούσαμε προηγουμένως. Ε, η ομάδα αυτή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα καθόλου το έτος και υπάρχουν και τεχνικοί εμπειρογνώμονες, ε, εργαζόμενοι του κλάδου δηλαδή, που συνεδριάζουν δύο με τρεις φορές το χρόνο. Ε, το πλαίσιο για τη δέουσα επιμέλεια ανανεώνεται συνεχώς. Τώρα έχουμε μια ενημερωμένη έκδοση του 2012 που θα τροποποιηθεί και πάλι και θα ενημερωθεί. Στόχος της κοινή προσέγγισης είναι να έχουμε ίσους κανόνες παιχνιδιού παντού σε όλες τις χώρες του ΩΣΑ και στους ε, ε, αντίστοιχους φορείς και να υπάρχει μια ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών ε, όσων καλούνται να εφαρμόσουν την κοινή αυτή προσέγγιση. Η κοινή προσέγγιση αναφέρεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες προδιαγραφές και πρότυπα, ιδιαίτερα της Παγκόσμιας Τράπεζας, που χρησιμοποιούν και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ακόμα και εμπορικές τράπεζες, ε, με βάση τις δικές τους ε, αρχές. Είναι benchmark, δηλαδή συγκριτική αξιολόγηση στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Όλα αυτά με φέρνουν ε, στο εξής σχόλιο. Η μελέτη αντικτύπου ως προς το περιβαλλοντικό και το κοινωνικό σκέλος σήμερα είναι πλήρως ενταγμένη στις δραστηριότητες ενός φορέα εξαγωγικών πιστώσεων, της αρχής μάλλον εξαγωγικών δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι εταιρείε που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε χώρε του ΟΣΑ βρίσκονται σε πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Όλο και περισσότερο έρχεται ανταγωνισμό από χώρε εκτό ΟΣΑ, π.χ. Κίνα. Οπότε είναι πάρα πολύ κρίσιμο να έχουμε υπόψη μας το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στα δικά μας σχετικά υψηλά πρότυπα ε, και για χώρες ε, του ΩΣΑ και τις αντιστοιχές αρχές των εξαγωγών και άλλες χώρες που έχουν πιο χαλαρά πρότυπα, δεσμεύσεις και προδιαγραφές. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε ίσους κανόνες παιχνιδιού ε, παγκοσμίω και όχι μόνο σε χώρες του ΩΣΑ. Π.χ. η γερμανική κυβέρνηση υποστηρίζει την πρόοδο της Διεθνούς Ομάδας Εργασίας ακριβώς έτσι ώστε να επεκταθούν οι συζητήσεις και σε εγκάρσια θέματα ή οριζόντια όπως είναι κοινωνικά, περιβαλλοντικά κτλ. Sorry. This way around. Um, just, uh, this slide... Αυτή η διαφάνεια εδώ σας δείχνει κάποια στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην δέουσα επιμέλεια ε, για τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να τονίσω ένα ζήτημα που στην πράξη παίζει σημαντικό ρόλο. Σύμφωνα με τις κοινέ προσεγγίσεις, ε, ο φορέας που διέπει τις εξαγωγικές πιστώσεις δεν θα πρέπει να κοιτάζει μόνο τα τεχνικά, ας πούμε, τον εξοπλισμό, τον τεχνολογικό, αλλά θα πρέπει να εξετάζει όλο το έργο επιτόπου, ας πούμε, θέλει κάποιος να χτίσει ένα πετροχημικό εργοστάσιο. Ε, συχνά έχει να κάνει με τη μόχλευση και με την επιρροή και των εξαγωγέων και του φορέα ε, που εποπτεύει τις εξαγωγικές πιστώσεις. Ε, θα πρέπει λοιπόν να εξετάζονται εκεί και τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά ζητήματα και όχι μόνο το οικονομικό σκέλος. come briefly to Uh, Έρχομαι τώρα στη διαφάνεια, άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα. Ο David Drysdale επίσης ε, αναφέρθηκε σε αυτό. Ε, τι κάνουμε ήδη και τι πρέπει να κάνουμε. Η κοινή προσέγγιση του ΩΣΑ σήμερα απαιτεί υψηλό επίπεδο διαφάνειας. Εκ των προτέρων θα πρέπει να δημοσιεύονται τα στοιχεία και να υπάρχει ενημέρωση για έργα της λεγόμενης κατηγορίας Α που ε, έχουν ε, ενδεχομένως υψηλό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Τι εννοώ κοινωνικό, κατεξοχήν εδώ εντάσσονται και εξορισμού τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όταν έχουμε ένα έργο κατηγορίας Α, οι ε, φορείς εξαγωγικών πιστός θα πρέπει να δημοσιεύουν τα στοιχεία 30 μέρες πριν την τελική δέσμευση και τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά και στη συνέχεια όλα τα έργα κατηγορίας Α και Β θα πρέπει και εκ των υστέρων να κοινοποιούνται στον ΩΣΑ εφόσον έχει δοθεί η κάλυψη από το φορέα μας. Υπάρχει και άλλος τρόπος για να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και γενικότερα στην πολιτική και στο συγκεκριμένο έργο κάθε φορά και σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΩΣΑ. Και έρχομαι στην τελευταία σύντομη διαφάνεια για να σας δώσω έτσι μια ιδέα για το πώς τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά στοιχεία ενός έργου ε, λαμβάνονται υπόψη στην Euler Hermes στη Γερμανία όταν καλύπτουμε τις εξαγωγικές πιστώσεις. Έχουμε μια διεπιστημονική ομάδα επιστημόνων, ε, ε, εμπειρογνωμόνων σε διάφορα επίπεδα, 11 υπαλλήλους, η αηφορία, και η βιωσιμότητα είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας αξιολόγησης και πολλές φορές είναι και ε, ένα θέμα που συζητείται σε μια διυπουργική επιτροπή. Η δέουσα επιμέλεια είναι κοινή στον όσα δεν θα σας εκπλήξει και επίσης γίνεται αναφορά σε διεθνείς προδιαγραφές ή πρότυπα συν ενδεχομένως συμπληρωματικές εθνικές διατάξεις όταν υπάρχουν η γερμανική προσέγγιση ε, έχει το εξή χαρακτηριστικό. Απόφαση παίρνουν τέσσερα υπουργεία και μάλιστα ομόφωνα καλούνται να λάβουν την απόφαση. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν ε, είναι αξιοσημείωτο ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ε, προσέχουν πάρα πολύ τα κοινωνικά θέματα, τα ανεπτυξιακά και τα περιβαλλοντικά. Ολοκληρώνεται εδώ η παρουσίαση μου και με χαρά να απαντήσω συνέχεια σε τυχόν ερωτήσεις που θα έχετε. Ευχαριστώ πολύ και τελευταίος τώρα ομιλητής από τους εμπειρογνώμονους είναι ο κύριος Παόλο Γκρατσότη, επικεφαλής ε, τμήματάρχης από την Γενική Διεύθυνση ε, εμπόριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιος για θέματα συντονισμού του ΠΟΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο που μας έδωσε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το σημαντικό θέμα. Ιδιάζον ε, θέμα για την εμπορική πολιτική, γιατί η εμπορική πολιτική είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράλληλα όμως δεν έχουμε μια τέτοια ευρωπαϊκή εξαγωγική υπηρεσία. Βασιζόμαστε δηλαδή στην εμπειρογνωμοσύνη και πραγματογνωμοσύνη των κρατών μελών διαπραγματεύοντας τους κανόνες και στην πολιτική καθοδήγηση αυτών. Τρεις εκθέσεις πρέπει να σας δώσουμε, να σας δίνουμε κάθε χρόνο, με βάση τον κανονισμό του 2011 33 τις ετήσιες δραστηριότητες όλων των κρατών μελών και με βάση αυτές η Κομισιόν δίνει μία επισκόπηση στο Κοινοβούλιο κάτι που κάνουν, τη δουλειά που κάνει την ετοιμάζει η Κομισιόν και μετά κάνει μια έκθεση για τις ε, διαπραγματευθήσεις δραστηριότητε. Έχουμε καθυστερήσει με αυτή την έκθεση, αλλά υπάρχουν ε, εξελίξεις στην ε, διεθνή ομάδα ε, που θέλουμε να τις ε, ε, εντάξουμε. Για τις τρεις πτυχές που αναφέρθηκαν οι προηγούμενοι ομιλητές, ε, όσα, κυρίως το arrangement, η συμφωνία, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέρος. Είδαμε το ιστορικό αυτής της συμφωνίας, ήταν επιτυχής, ήταν, ήταν αποτελεσματικό ε, εργαλείο για να εξασφαλίσει την ισοτιμία στα προγράμματα εξαγωγικών πιστώσεων. Ε, δεν υπάρχει επιδότηση στη χρηματοδότηση των ε, εξαγόμενων αγαθών και η Βραζιλία αποφάσισε, επειδή ακριβώς ήταν τόσο επιτυχές, να ενταχθεί σε αυτό το arrangement, ενώ δεν εμπλέκεται και δεν συμμετέχει στον όσα Φυσικά, ε, οι εξαγωγικέ πιστώσει είναι εμπορικό εργαλείο. Ε, η δέουσα επιμέλεια, όμω, όταν εξετάσουμε τα προγράμματα, είναι βασικό στοιχείο, όπω ακούσαμε από τον Οργανισμό Εξαγωνικών Πιστώσεων. Υπάρχει μια νέα αναθεώρηση των κοινών ε, προσεγγίσεων για την ε, κοινωνική και περιβαλλοντική ε, δέους επιμέλεια, ούτω ώστε να αναπτύξουμε την διάσταση που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και σημειώσαμε το ψήφισμα του Κοινοβουλίου για το πώς η μεθοδολογία για τη δέουσα επιμέλεια μπορεί να βελτιωθεί στις εξαγωγικές πιστώσεις. Ο ΣΑ είναι το μοναδικό, ο μοναδικός φορέας που έχει πραγματογνωμοσύνη. Πιστεύουμε λοιπόν ότι οι συζητήσεις που γίνονται εκεί μπορεί να αποτελέσουν τη βάση για το δικό μας προβληματισμό. Τώρα, αν δεν αρκεί αυτά που λέει όσα για να δεσμευτούν όλοι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων, μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάποια ευρωπαϊκά πρότυπα. Όπως είπε και ο κύριος ε, Γιούγκερ, στις εξαγωγικές πιστώσεις ε, πέρα από τον ΩΣΑ αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη πρόκληση. Η συμφωνία του ΩΣΑ ήταν αποτελεσματική, όπως είπαμε. Ε, αλλά έχουμε νέους παρόχους εξαγωγικών πιστώσεων τα τελευταία χρόνια που προέκυψαν και δεν ανήκουν στον ΩΣΑ και δεν δεσμεύονται από το arrangement του ΩΣΑ. Κίνα, Φερρυπίν. Αλλά και Ινδία, Βραζιλία, Νότιο Αφρική και, και Ρωσία βέβαια. Το πώ θα εμπλέξουμε αυτές τις χώρες είναι η μεγάλη πρόκληση σε εξαγωγικέ πιστώσεις τον 21ο αιώνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΠΑ και άλλοι συμμετέχοντα του ΩΣΑ το συζητάνε με την Κίνα, τη Βραζιλία, την Νότια Αφρική, την Ινδονησία και άλλους και άλλους ε, αναδυόμενους παρόχους εξαγωγικών πιστώσεων. Θα σας πούμε περισσότερα στην έκθεση που ετοιμάζουμε. Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε πριν από χρόνια, το 2011, αν θυμάμαι καλά, με τον αντιπρόεδρο της ε, Κίνας και τον πρόεδρο Ομπάμα. Ο στόχος ήταν να φτάσουμε σε συμφωνία μέχρι το τέλος του 2014. Με δυσκολία ξεκίνησε, όπου συζητήσαμε ε, το ιατρικό εξοπλισμό και τα πλοία, εκεί τις εξαγωγικές πιστώσεις, δηλαδή σε αυτούς τους τομείς. Ε, πριν από πολλές εβδομάδες ε, συναντηθήκαμε με την Βραζιλία, τώρα ε, θα συζητήσουμε και καθολική, καθολικά με την Κίνα, για όλους τους τομείς δηλαδή. Είναι μεγάλη η πρόοδος για μας και θα εφαρμόσουμε τη μετάβαση στη νέα φάση στο IWG. Το ECA Watch είπε στην αρχή ότι γίνονται σημαντικές συζητήσεις για τις εργατικές πιστώσεις και την επίπτωση στο, στην κλιματική αλλαγή λόγω της πολιτικής εστίασης στο G7 που υπάρχει στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Ειδικά για τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν τον άνθρακα. Θέλουμε εμείς να είμαστε έτοιμοι εγκαίρως για αυτό το θέμα ε, εν ώψη του, COP, του COP21 παρότι είναι πολύ δύσκολο θέμα και πολύ αμφιλεγόμενο και στον ΩΣΑ και στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο νέος πρόεδρος της ομάδας του ΩΣΑ υπεύθυνο για τις διαπραγματεύσεις ε, ξεκίνησε, υπέβαλε μια νέα πρόταση που κατά την άποψή μας ε, είναι λογική βάση για να επιτευχθεί συμβιβασμό. Η, η Κομισιόν ετοιμάζει μια πρόταση προς το Συμβούλιο με βάση το άρθρο 29 της Συνθήκης για ε, τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια νέα θέση ε, για αυτή την πρόταση του ΩΣΑ και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να διευκολύνουμε μια επικοδομητική λύση μέχρι το COP21 για τις εκθέσεις τώρα που λαμβάνεται, Ακούσαμε και κάποιες προτάσεις από την ΕΣΥΑ για το πώς θα τις βελτιώσουμε. Περιμένουμε να ακούσουμε τις προτάσεις σας ε, για το πώς θα βελτιώσουμε αυτές τις εκθέσεις. Φυσικά Κάποια πράγματα μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά κάποια άλλα όμως έχουν να κάνουν με τη συμφωνία που επετέφθη το 2001. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε από πλευρά Επιτροπή, Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με βάση την πολιτική συμφωνία και με βάση το arrangement, τη συμφωνία του ΟΣΑ, δηλαδή δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση μονομερώς να αλλάξουμε τις παραμέτρους ε, της συμφωνίας. Φυσικά ε, περιμένουμε την καθοδήγησή σας και την τεχνική υποστήριξη από τα κράτη-μέλη για να βελτιώσουμε τη δουλειά που κάνουμε στον ΩΣΑ, που παραμένει ακόμα και σήμερα ο μοναδικός φορέας και θεσμός ε, και το μόνο νομικό πλαίσιο για να μας δώσει για, να, για τις εξαγωγικές πιστώσεις. Ε, η μόνη ε, δυνατότητα για να ενισχύσουμε και το arrangement αλλά και την ε, μεθοδολογία για την δέουσα επιμέλεια. Και κάνουμε ε, ό,τι μπορούμε για να πετύχουμε μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα καλύτερο αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις. Γιατί σήμερα το να έχουμε ένα κλαμπ από αναπτυγμένες οικονομίες με κοινού κανόνες για τις εξαγωγικές πιστώσεις και εκτός του κλαμπ παίχτες όπως εκείνα που δεν έχει την ίδια προσέγγιση και δεν ακολουθεί τους ίδιους κανόνες. Είναι δύσκολο, είναι μια πρόκληση που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση, Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ πρώτα ε, ο εισηγητής και μετά ο κύριος Φίσας. Ε, Γιάννη Σας ευχαριστώ. Την πρώτη φορά που είχαμε συζητήσει στην Επιτροπή Εμπορίου Διεθνούς Εμπορίου αυτό το θέμα Είχαμε ακούσει τον εκπρόσωπο του ΟΣΑ και τον εκπρόσωπο του Ερμές, του Hermes, που έλεγαν πάνω κάτω αυτά που ακούσαμε και σήμερα. Δηλαδή, από την πλευρά του ΟΣΑ λέει εργαζόμαστε, προσπαθούμε να προχωρήσουμε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κοινέ στρατηγικές, αλλά αυτό παραμένει και πρέπει να παραμείνει για να γίνεται στο επίπεδο του ΟΣΑ. το οποίο σημαίνει ότι συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως, ως οργανισμός εκεί, αλλά πρώτα απ' όλα το έργο γίνεται στο επίπεδο των κρατών μελών. Εξετάζοντας το θέμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάλαβε γρήγορα ότι το ζήτημα αναφέρεται, έχει σχέση μάλλον με την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις εξωτερικές της σχέσεις, επομένως πρέπει να ανταποκρίνεται και στην πολιτική μας για το θέμα αυτό και στις ε, προβλέψεις της συνθήκης για το θέμα αυτό και έτσι καταλήξαμε σε, στην ανάγκη να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός λογοδοσίας και παρακολούθησης του τι γίνεται στο επίπεδο των κρατών μελών. Και καταλήξαμε σε μια συμφωνία, σύμφωνα με την οποία τα κράτη-μέλη οφείλουν να συμφωνούν ε, και να ακολουθούν και να προωθούν τους στόχους της συνθήκης, κατά πρώτον. Κατά δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να επεμβαίνει, να ασκεί πίεση στα κράτη-μέλη, να βοηθά από πλευρά μεθοδολογικής και να λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μετά από πάρα το 2-3 ετών καταλήξαμε σε ένα σύστημα το οποίο διασφαλίζει αυτή τη λογοδοσία και διασφαλίζει ότι αυτή η μεθοδολογία όχι απλώς υπάρχει, αλλά εφαρμόζεται κιόλα. Γιατί δεν αρκεί, όπως ακούσαμε από τον εκπρόσωπο του, εκπρόσωπο του Ερμές, ε, να λέμε μην ανησυχείτε, λαμβάνουμε υπόψη μας τα θέματα του περιβάλλοντος. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ε, μια λογοδοσία, να γνωρίζουμε ακριβώς ε, πώς, πώς μετράτε η επίπτωση στο περιβάλλον όταν παρέχουμε αυτές τις εξαγωγικές πιστώσεις ή όταν χρηματοδοτούμε κάποια διεθνή project, κάποια διεθνή έργα σε διεθνές επίπεδο. Έχουν περάσει λοιπόν τρία-τέσσερα χρόνια και μπορούμε πλέον να αξιολογήσουμε ε, την ποιότητα των εκθέσεων που υποβάλλουν οι οργανισμοί ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων και η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διαπιστώνουμε ότι παραμένει χαμηλή αυτή η ποιότητα. Δεν έχουμε ξεπεράσει τις αναφορές στο έργο που γίνεται στο επίπεδο του ΟΣΑ. Δεν αναφερόμαστε όσο θα έπρεπε στο τι γίνεται στα κράτη-μέλη και στο επίπεδο της Ένωσης. Και με άλλα λόγια, απλώς ακούμε τους οργανισμούς στα, εθνικά, στα κράτη-μέλη να μας λένε ότι βασικά δεν είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, είναι αυτοί οι οργανισμοί ε, ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων που χρηματοδοτούν στο μεγαλύτερο βαθμό παγκοσμίω τα ε, ορυκτά καύσιμα και τον άνθρακα. Αυτό αντακατοπτρίζει την πολιτική μα ως Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έλεγα πω όχι. Από την πλευρά τη Επιτροπής ακούμε, ναι, θα προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε, να κάνουμε κάτι παραπάνω, αλλά ε, όχι και πολλά. Επομένω, η Επιτροπή Διεθνού Εμπειρίου πρέπει να ε, σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά εάν θέλει να αναθεωρήσει ή να επανασυμφωνήσει ε, στις... Ε, ο κύριος Φύσης, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της Κίνας, γιατί έγινε μεγάλη κουβέντα. Είναι αρκετά ανησυχητικό αυτό το θέμα. Ε, ασχολείται πολύ με την Αφρική και πριν από ε, λίγα χρόνια υπήρχε μια εκλογική αντιπροσωπεία ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον Νίγηρα, όπου φτιάχναν ένα, ένα σημαντικό, μια σημαντική γέφυρα στο ποταμό ε, και υπήρχε και ένα πετροχημικό εργοστάσιο με κινέζικες ε, Όταν εγώ μίλησα με τους υπουργούς και με την κυβέρνηση του Νίγηρα, πώς γίνονται όλες αυτές οι επενδύσεις πώς εμπλέκεται η Κίνα, η οποία ε, στην πραγματικότητα δεν χρησιμοποιεί τον τόπιο εργατικό δυναμικό. Φτιάχνει, ας πούμε, κάτι εκεί ξεν, έτσι, ξενώνες, ξέρω εγώ, φέρνει κόσμο απ' έξω, δεν χρησιμοποιεί ντόπιου. Οι Κινέζοι δεν είναι αυστηροί και νομίζω ότι υπάρχει θέμα του ανταγωνισμού για αυτές τις εταιρείε, για αυτούς τους ε, εργαζόμενους πρέπει να υπάρξουν ε, ριζικά μέτρα και αποτελεσματικά μέτρα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εμείς είμαστε οι πρώτοι δωρητές αναπτυξιακής βοήθειας, αλλά δεν θα μπορούμε σε καμία περίπτωση να υλοποιούμε αυτά τα έργα, ε, ενώ είμαστε απόλυτα λογικοί στους όρους που θέτουμε εμείς, ενώ οι Κινέζοι δεν είναι με ποια συγκεκριμένη μορφή μπορούμε να αποφύγουμε το πρόβλημα αυτό που δημιουργούν οι Κινέζοι. Ναι, ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Έχω μια ερώτηση ίσως από άγνοια και ζητώ συγγνώμη που δεν το γνωρίζω, αλλά ε, έχετε εστιάσει πολύ στην πλευρά της προστασίας του περιβάλλοντος που συμφωνώ είναι πάρα πολύ σημαντική ε, όταν μιλούμε για αυτούς τους τομείς. Αλλά φαίνεται ότι η κοινωνική διάσταση ανάγεται ε, αποκλειστικά στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και εγώ δεν έχω καταλάβει τι περιλαμβάνεται εκεί, εργατικά δικαιώματα, εργασιακά ζητήματα, κοινωνική κοινωνικής προστασίας γενικότερα ε, και εφαρμογή της νομοθεσίας θα μπορούσατε να μας απαντήσετε λίγο περισσότερα για το τι συμπεριλαμβάνεται στη δέουσα επιμέλεια ως προς κοινωνικά κριτήρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει άλλος που να έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλούνται οι εμπειρογνώμονες για να απαντήσουν σύντομα έκαστος. Ο κύριος Ντάιστελ. Ε, Yes, thank you. Um, in the context of the common approaches... Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τον... τη συμφωνία πλαίσιο που είναι η κοινή προσέγγιση του ΩΣΑ, εδώ είναι μια συμφωνία στην οποία τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στο ΩΣΑ έχουν συμφωνήσει να εφαρμόζουν τα διεθνή πρότυπα, τα οποία ποικίλουν. Γιατί ω γνωστό δεν είναι συνεκτικά τα ίδια μεταξύ του τα διεθνή πρότυπα. Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά ε, πρότυπα. σε ορισμένα ε, συμπεριλαμβάνονται για παράδειγμα τα εργατικά δικαιώματα. Ενώ σε άλλα προγράμματα, αν για, αν για παράδειγμα χρηματοδοτείται ένα έργο στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωση, θα εφαρμόζονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τα εργατικά δικαιώματα. Που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα εξαρτώνται όλα από την χώρα στην οποία θα υλοποιηθεί το έργο και αν Να σας δώσω ένα ε, τυπικό παράδειγμα. Εάν απλώς χρηματοδοτείτε 10 φορτηγά που θα χρησιμοποιηθούν για ένα έργο δισεκατομμυρίων, δεν έχετε και πολλά να πείτε για τα πρότυπα που θα εφαρμοστούν. Εάν δίνετε 2 από τα 10 δισεκατομμύρια, θα σας ακούσουν περισσότερο σε σχέση με τα πρότυπα που θα εφαρμόσουν. Τα μέλη μας, πάντως, ακολουθούν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις ε, συνδυασμού αυτών των διεθνών προτύπων. Ορισμένε φορέ συμπεριλαμβάνονται και τα εργατικά δικαιώματα στα ανθρώπινα δικαιώματα, άλλοτε όχι. Μήπω μπορείτε να απαντήσετε και στο ερώτημα του κυρίου Φίσα για αυτόν τον ανταγωνισμό μεταξύ των κινέζικων επενδύσεων και των ε, επενδύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τι επιπτώσει έχει αυτό στα πρότυπα. Απάντηση. Δύσκολο είναι πάντα να κρίνουμε αυτό που κάνει ή δεν κάνει η Κίνα γιατί δεν υπάρχει δημοσιότητα, δεν υπάρχει διαφάνεια στις ενεργειές της. Γι' αυτό από την πλευρά του ο ΣΑ προσπαθεί να δημοσιοποιεί τις ενεργειές του και να υπάρχει λογοδοσία και διαφάνεια. Για να είναι ξεκάθαρος ποιες πολιτικές προωθούνται με τις ενέργειές μας. Προσπαθούν μέσω της Διεθνούς Ομάδας Εργασίας οι Ηνωμένες να πιέσουν την Κίνα να ανοιχτεί περισσότερο και να συμμετάσχει περισσότερο όπως έχουν δεσμευτεί και τα μέλη του ΩΣΑ, άλλες 18 χώρες που δεν είναι μέλη του ΩΣΑ και συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα. Ε, βεβαίως αυτή η διαδικασία είναι πολύ αργή, γιατί τα μέλη του ΩΣΑ έχουν ήδη ένα πολύ καλά αναπτυγμένο σύστημα, το οποίο συμπεριλαμβάνει και τις βέλτιστες πρακτικές για τη διακυβέρνηση το οποίο δεν το αγγίζει καν η συζήτηση στη Διεθνή Ομάδα Εργασία. Το μόνο που συζητάτε αυτή τη στιγμή είναι η όρη χρηματοδότηση στη Διεθνή Ομάδα Εργασία. Επομένω, δεν γνωρίζουμε πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα δούμε. Πάντω, η Κίνα προσπαθεί να κερδίσει έδαφο, προσπαθεί να συμμετάσχει στην IWG, στην Διεθνή Ομάδα Εργασία, αλλά αυτό συμβαίνει αργά και πρέπει να γίνει μεθοδικά. Πάντω, όλοι φαντάζομαι επιθυμούν να δημιουργηθεί ένα συσότιμο ανταγωνισμό και έτσι ώστε οι χρηματοδοτήσει από τι διάφορε κυβερνήσει να μην στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Θα δείξει, θα όμω τι θα συμβεί στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριο Πάρα πολύ σύντομα για τα κοινωνικά ζητήματα. Νομίζω εν μέρη έχουν ληφθεί υπόψη Ε, στην αρχή ήταν πολύ στενό το περιβαλλοντικό πλαίσιο, ε, δεκτείνεται σε κοινωνικό. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουμε μεγάλους περιορισμούς, δεν έχουν οριστικοποιηθεί αυτά. Για τα ε, εργασιακά δικαιώματα κάποιες φορές συμπεριλαμβάνονται και κάποιες φορές αλλού ε, υπάρχουν ε, φαινόμενα όπως και στην Ινδία παιδικής εργασίας. Αυτή τη στιγμή έχει ένα σύστημα εγκαθιδρυθεί, εγκατασταθεί, δεν αλλάζει πολύ εύκολα. Ε, και ειδικά στην αλυσίδα παροχής για, την Κίνα, να πάρω ένα παράδειγμα για τον άνθρακα. Η κινέζικη κυβέρνηση όπως και η Ιαπωνική και η Κορεατική που είναι στον ΩΣΑ υποστηρίζουν τον άνθρακα και τεχνολογίες και αντιπαραγωγικές και, και παραγωγικές. Εμείς θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει κρατική ενίσχυση καθόλου για τον άνθρακα. Αλλά η κατάσταση είναι ανάμεικτη. Επειδή ενδιαφέρονται ε, οι Κινέζοι να μπουν και στο παγκόσμιο σκηνικό, πρέπει να δούμε πώς θα δώσουμε εμείς το καλό παράδειγμα, οι δικές μας κυβερνήσεις. Υπάρχει μια στεναρή αντίσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γερμανίας γιατί χρειάζεται περισσότερη φιλοδοξία όπως το είπε και ο πρόεδρος Ολάντ και κάποιοι άλλοι. Νομίζω λοιπόν ότι θα κριθούμε εκ του αποτελέσματος και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σε χώρες ΩΣΑ, μη και να επιτευχθεί περισσότερη πρόοδος επί τόπου. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ε, προσθέσω κάτι σε αυτό που είπε ο David Drysdale. Ε, τι γίνεται με τις προδιαγραφές που χρησιμοποιούμε το IFC, ε, που χρησιμοποιούν και το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο. Έχει κάνει αυτή η Επιτροπή IFC μελέτες στο παρελθόν για να δει ε, που υπάρχουν ε, ρογμές ή διαφορές ανάμεσα στα διάφορα προγράμματα, στα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει δείκτες λοιπόν επιδόσεων ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης που έχουμε και εμείς συμπεριλάβει. Πάντα όμως δεν υπάρχει πάντα η επικεφαλίδα ή ταμπέλα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, είναι σε ένα επίπεδο ειδήσει όπου πολλά από τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται υπόψη χωρίς πάντα να αναφέρονται ρητά ε, ούτε να μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι 100% ε, τα τηρεί αυτά το έργο. Μα εδώ έρχεται και ο ρόλος του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Επιστώσεων της κάθε χώρας για να ελέγχει, να εποπτεύει το έργο. Καμιά φορά έχουμε και εξωτερικούς συμβούλους που ε, υπησέρχονται. Εξαρτάται αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό από το κάθε έργο κάθε φορά. Ευχαριστώ κύριος ε, ε, Γκαρτσότη. Ευχαριστώ. Δεν θα μπω εγώ στο θέμα των κοινωνικών δικαιωμάτων και των προτύπων. Το εκάλυψαν οι προλαλήσαντες. Εγώ θα σταθώ στο ζήτημα της Κίνας και το πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει παράδειγμα. Γιατί πράγματι ο άνθρακας είναι ένα καλό ε, παράδειγμα. Τι είναι οι εξαγωγικές πιστώσεις. Είναι ένας μηχανισμός για να βοηθήσει τις εταιρείε να εξάγουν προς περιοχές του κόσμου όπου οι πιστώσεις, ε, το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν είναι εξίσου αξιόπιστο ή εύκολο. Επομένως, θέλουμε τα δημόσια χρήματα που θα επενδυθούν, που θα δοθούν με τη μορφή πιστώσεων με αυτόν τον τρόπο, να γίνει με τε αυτό με τρόπο συμβατό προς τις αρχές μας και ταυτόχρονα να μην στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός στις ε, ε, εξαγωγές. Και αν θέλετε αυτό που ζητάτε από την Κομισιόν είναι να τετραγωνίσει τον κύκλο που δεν είναι εύκολο και σας θέτω πιο συγκεκριμένο το ερώτημα. Εμείς ως ε, μέλη του ΟΣΑ έχουμε μια πιο φιλόδοξη θέση όσον αφορά στο κατά πόσο πρέπει να χρησιμοποιείται ο άνθρακας κτλ. Επομένως, εάν εμείς αποσύρουμε τις χρηματοδοτήσεις μας σε αυτά τα προγράμματα, θα, καλύψει το κενό, θα καλύψουν το κενό χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, το Βιετνάμ, που έχει χαμηλότερα πρότυπα. Επομένως, αυτό πρέπει να κάνουμε ή να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε έτσι ώστε μέσω της χρηματοδότησης να πιέσουμε για την υιοθέτηση ψηλότερων προτύπων ε, κατά πολέμηση κλιματική αλλαγής. Αυτό δεν θα σας δώσω εγώ την απάντηση, πάντως από την εμπειρία μου έχω διαπιστώσει ότι αυτή δεν είναι μια κατάσταση ε, όπου είτε, είτε άσπρο είτε μαύρο. Δεν είναι... Πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση και γι' αυτό είναι και χρήσιμος ο διάλογος που κάνουμε σήμερα. Και γι' αυτό είναι, έχει και αξία εξάλλου η λογοδοσία της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο. Και μια διευκρίνηση δεν είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνουμε ό,τι μπορούμε με αυτό που έχουμε. Εξαντλούμε τα περιθώρια του θεσμικού μας ρόλου. Βεβαίως με τους περιορισμούς που ε, δεν μπορούμε μερικές φορές να ελέγξουμε. Για παράδειγμα, αν δεν υπάρχει λογοδοσία και δημοσιότητα στην ε, πηγή, πώς μπορούμε να έχουμε εμείς τα δεδομένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους εμπειρογνώμονες και τους συναδέλφους που μίλησαν μας δώσατε πολύτιμα στοιχεία τα οποία θα τα συμπεριλάβουμε στις εργασίες μας και θα τα συζητήσουμε για τις κατεξουδότηση πράξεις μετά το καλοκαίρι για να υπάρξει και μια συνοχή και μια συνάφεια ε, στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουμε μια εξαγωγική πολιτική που να βασίζεται σε αρχές και αξίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ολοκληρώνεται αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης μαζί με τη δημόσια συνεδρίασή μας. Ραντεβού στις 4.30 για τη συνεδρίαση των συντονιστών. Σας ευχαριστώ πολύ.